άλλοι παράγοντε, γιατί δεν είναι μόνο οι συντάξει που επιβαρύνουν τα έλλειμματα, αυτό είναι λογικό. Και καθώ οδεύουμε προ την ιδέα συνολικών λύσεων, δεν μπορούμε συνεχώ να προβλέπουμε εξαιρέσει. Uh, thank you.